χρησιμοποιώντας και αυτή τη συμφωνία με αποτελεσματικό τρόπο και με σωστή διαχείριση. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να εμπλέξουμε τη Συμφωνία του Παρισιού και να προσφέρουμε και τις ευρωπαϊκές πράσινες λύσεις ε, σε όλο τον κόσμο. Πρέπει να αφήσουμε λοιπόν τα πολιτικά παιχνίδια και τα ταχυδικτυλουργικά Ευχαριστώ, κυρία Κέιτο, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Οι Ευρωπαίοι διαπραγματεύτε στις ε, συζητήσεις για το κλίμα θεωρούν ότι είναι ηγέτες ε, στην κλιματική αλλαγή, όμως ακόμα αγνοούν την επιστήμη και δεν λένε την αλήθεια για το κλίμα. Η αλήθεια είναι ότι θέλουμε καθαρά μηδενικέ εκπομπέ μέχρι το 2030. Αυτό είναι ριζικός τρόπος αλλαγής του τρόπου ζωή μα. Όταν επικεντρωνόμαστε στενά στις δικές μας άμεσες εκπομπές ε, αερίων, όμως δεν κοιτάμε τι γίνεται με τις εκπομπές διεξουδίου του άνθρακα σε αυτά που εισάγουμε, δεν έχει νόημα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν δεν θα έχει κανένα αποτέλεσμα αν δεν έχει διαφωτισμένη πολιτική. Πρέπει να έχουμε λοιπόν ε, στο μυαλό μας ότι έτσι δίνουμε το πράσινο φως για να καταστρέφεται ο Αμαζόνιος και να χάνουν την αιστεία τους ε, οι γηγενείς. Θέλουμε λοιπόν ε, μια φωτισμένη πολιτική και για τη δική μας Ήπειρο αλλά και για τους υπόλοιπους γιατί το περιβάλλον είναι ένα κοινό αγαθό για όλη την ανθρωπότητα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Χακαράινεν για δύο λεπτά. Και αυτό το θέμα έρχεται στην ημερήσια διάταξη μετά από πρωτοβουλία των Πρασίνων. Ε, πραγματικά πλανάστε να θεωρείτε ότι ε, αυτή η πίεση για το κλίμα θα έχει κάποιο αποτέλεσμα. Προσπαθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να θέσει στόχους για το κλίμα. Λέει για φόρους για το κλίμα, όμως ε, στέλνουν χρήματα ε, χωρίς ε, να υπάρχει συγκεκριμένος στόχος. Η νέα πράσινη συμφωνία βασίζεται στην εθελούσια συμμετοχή. Αν δεν γίνουν όμως όλα υποχρεωτικά, δεν θα πετύχουμε τους στόχους μας. Οι χώρες της Μερκοσούρ Ε, θα πρέπει να τηρήσουν αυτή την ε, συμφωνία και πραγματικά με τις τοπικές κουλτούρες ε, θα είναι δύσκολο να συμβεβαστεί αυτό. Η ομιλία Ε, στην ουσία ε, κατέληξε με τα ίδια λόγια ότι ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα χάσει από όλα αυτά. Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να δώσει ξανά την ισχύ στα εθνικά κράτη. Εκεί θα πρέπει να καταλήξουμε το Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα είναι στην ίδια ομάδα με την Ευρωπαϊκή Ένωση και εύχομαι στους Βρετανούς κάθε επιτυχία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 Ευχαριστούμε ο κύριος Ζεχράντιλ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Η συζήτηση για τις εμπορικές μας συμφωνίες και γενικώ για το εμπόριο είναι μια συζήτηση που πάντοτε έχει ιδεολογικές χρειές και ε, παίρνει πολιτικές διαστάσεις. Ήδη από την περασμένη κοινοβουλευτική θητεία συνέβαινε αυτό και τώρα η κατάσταση χειροτερεύει. Προσφάτως υπήρξε η προσπάθεια να αναβάλουμε ή τουλάχιστον να μην περάσει η συμφωνία με το Βιετνάμ διότι υπήρχαν κατηγορίες ό,τι αφορά τα κλωστοϊφαντουργικά. Σε ό,τι αφορά τη συμφωνία με τον Μαρκοσούρ, δεν αρέσει στην αριστερά τη Ευρώπη η Βραζιλία του Μπολσονάρου. Μιλάνε για τι ποσοστώσει, γεωγραφικέ ενδείξει, σε σχέση με τη συμφωνία αυτή όλα έχουν σχέση με την εμπορική μα πολιτική. Όμω, εμεί μιλάμε για ανθρώπινα δικαιώματα, για περιβαλλοντικά πρότυπα και κανόνε για θέματα που αφορούν άλλους θεσμούς ε, και οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όχι όσους ασχολούνται με τις εμπορικές συμφωνίες και για την πράσινη συμφωνία και τον δρόμο που θέλουμε να ακολουθήσουμε εμείς σε αντίθεση με τους υπόλοιπους. Ως προς τα εμπορικά όμως θα βρεθούμε να κλείνουμε τα εμπορικά μας σύνορα και να εμποδίζουμε τις συναλλαγές μας σχεδόν με όλους. Θα πρέπει λοιπόν όταν μιλάμε για εμπόριο να παραμένουμε συγκεντρωμένοι στα θέματα του εμπορίου αυστηρός. Ευχαριστούμε για ένα λεπτό η κυρία Ματίας. Ευχαριστώ πρόεδρε. Είναι πραγματικά αξιοπερίεργο πως το Ευρωκοινοβούλιο δέχτηκε εδώ το φύλλαρχο Ροάνη και τους άλλους φιναλές του βραβείου Ζαχάροφ, τους προσπιστές ε, του τροπικού δάσους της Αμαζονίας, χθες μόλις, και λέμε τώρα κατά πόσο είναι συμφωνία Μερκοσούρ ε, είναι συμβατή με την Πράσινη Συμφωνία. Δεν είναι. Ε, ας δούμε το δάσος του Αμαζονίου και τι συμβαίνει εκεί. Εδώ έχουμε απλώς ένα πρόσχημα στη συζήτηση αυτή για να βρούμε ε, δικαιολογεί αίτια και να προωθήσουμε το εμπόριο. Αυτή η συμφωνία θα καταδικάσει σε θάνατο την περιοχή του Αμαζονίου και θα είναι και βραβείο για τον Μπολσονάρο. Θα το πούμε και μπράβο. Ε, είναι πραγματικά προσβολή για του ε, ηθαγενεί, του πληθυσμού, του τοπικού και του ακτιβιστέ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πρέπει να το πετάξουμε στα σκουπίδια αυτό το αυτή τη συμφωνία. Ο Μπολσονάρου ήδη έχει πει ότι θα αποσυρθεί από τι περιβαλλοντικέ συμφωνίε. Και τι λέμε τώρα εδώ, δεν θα έχουμε καμία συμφωνία των Παρισίων και ε, πρέπει να είμαστε πολύ εύπιστοι ή πολύ υποκριτέ για να νομίζουμε ότι όλα θα πάνε καλά. Εγώ είμαι από την πλευρά, ε, στο πλευρό των ακτιβιστών του Αμαζονίου και όχι των υποκριτών σε καμία περίπτωση. Ευχαριστούμε. Επόμενος για 1,5 λεπτό ο κύριος Σαλίνη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καλησπέρα Επίτροπε. Οι εμπορικές μας σχέσεις ε, με την Μερκοσούρ ξεπερνά τα 20 δις ευρώ ως προς την ανταλλαγή αγαθών και υπηρεσιών. Ένα σημαντικότατος όγκος ε, ως προς τη χρηματική αξία και όπως είπε προηγουμένως ο συνάδελφος Ζήμων, ε, σήμερα ήδη στο εμπορικό επίπεδο βλέπουμε να μην υπάρχει σεβασμός για τους βασικούς κανόνες Όπω θα έπρεπε να γίνεται. Ε, και συζητάμε τώρα τι προσδοκίες όλων μας ως προς την Πράσινη Συμφωνία. Ναι, αλλά εμένα αυτό που με ενδιαφέρει ιδιαίτερα είναι η ομάδα των Πρασίνων που θέλει να αντιδράσει τόσο συγκροτημένα ως προς το γεγονός ότι υπάρχει πρόεδρο ε, τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή που ανέλαβε να προωθήσει την πράσινη συμφωνία ε, με συνέπεια. Όμω εδώ δεν ε, φάνηκε να αντιδρούν λογικά. Δηλαδή ξεκινάνε να παίζουν ένα πολιτικό παιχνίδι λίγο επικίνδυνο ποιο θα κλωτσίσει την μπάλα μακρύτερα, ποιο θα φτάσει μακρύτερα. Δηλαδή, εδώ μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για πολιτική συμφωνία. Ε, ε, πράσινη συμφωνία, μάλλον. Συμφωνία σημαίνει ότι όλοι πρέπει να συμφωνήσουν. Μην γινόμαστε τώρα εδώ λιγότερο σοβαροί. Ε, Όλοι πρέπει να συμφωνήσουν και όλες οι εμπορικές συμφωνίες. Ε, με ε, παντιέρα το, την πράσινη συμφωνία θα πρέπει τώρα να αξιολογηθούν εκ νέου, διότι η πράσινη συμφωνία δεν θέλουμε να γίνει κινητήριος δύναμη όλης της Επίρου, αλλά να γίνει τα φόπλακα της Ευρώπης, δηλαδή ε, να μην μπορέσουμε να καταφέρουμε τίποτα με αυτή τη συμφωνία. Εμείς θέλουμε κάτι ε, τελείως διαφορετικό. Να εργαστούμε για τους πολίτες και το καλό τους, όχι για να πάρουμε τέσσερις ψήφους παραπάνω όπως κάνετε εσείς. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Διεντρών. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έχουμε ένα πολύ προβληματικό ντοσχέ μπροστά μας. Η συμφωνία αυτή είναι γραμμένη σε, με όρους ακατανόητους. Δεν καταλαβαίνουμε τι λέει διότι σήμερα ο κόσμος χρησιμοποιεί πλέον άλλο λεξιλόγιο. Έχουμε μπροστά μας ένα κουτί της Πανδώρας. Δημιουργήθηκε για τον κόσμο όπως ήταν πριν από 20 χρόνια και βασίστηκε στην πίστη ε, ότι ο κόσμος αυτός μπορεί ακόμα να υπάρχει. Όχι, η συμφωνία αυτή έχει ε, γραφτεί ε, με γνώμονα το χρήμα και στο, θυσιάζοντας το περιβάλλον, την κοινωνία και τις τοπικές κοινωνίες. Με τις πυρκαγιές στα τροπικά δάση και ε, τους των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεν μπορούμε να προσυπογράψουμε σε συμφωνία και να δεχτούμε αυτή την υποκριτική στάση. Οι πολίτες μας απαιτούν να διαμαρτυρόμαστε κατά τέτοιων συμφωνιών. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας. Για τη συμφωνία αυτή και για να μεταφραστεί σε μια σύγχρονη γλώσσα, γλώσσα που ακόμη δεν υπάρχει, που να περιλαμβάνει τα ανθρώπινα δικαιώματα και την περιβαλλοντική προστασία, ε, ο κόσμο βγαίνει στου δρόμου και το απαιτεί αυτό, το διεκδικεί. Εμεί δεν μπορούμε με γεμάτη χαρά να δίνουμε βραβεία για την ειρήνη και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ταυτόχρονα να απαρνούμαστε τα θεμελιώδη δικαιώματά μα για να πάρουμε περισσότερα κινητά και αυτοκίνητα. Ευχαριστούμε. Η κυρία Μπιλμπάου, για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ. Η Πράσινη Συμφωνία στο σημείο 3 αναφέρεται στο ότι η Ένωση θα πρέπει να γίνει παγκόσμιος ηγέτη στην οικολογική μετάβαση. Ένα από τα εργαλεία είναι η εμπορική πολιτική. Η συμφωνία με τη Μερκοσούρ περνάει από τα λόγια στα έργα. Μετά τη Συμφωνία των Παρεσιών είναι απέτηση αυτό και στο μέλλον θα γίνει. Έχει δώσει ήδη καρπούς αυτή η ρήτρα. Νομίζω ότι οδήγησε στο σύμφωνο της Λετήσια για την Αμαζονία ως ε, απάντηση στις δασικές πυρκαγιέ. Γι' αυτό ε, πιστεύω ότι θα ε, συνεχίσουμε στο σωστό δρόμο και χαίρομαι και το χειροκροτώ αυτό. Έχουμε πολύ μεγάλη ευθύνη για την βιωσιμότητα και η φορεία. Και τέλος, ελπίζω πολύ στο ότι θα πρωταγωνιστήσουν οι πολίτε. Σήμερα συζητούμε γιατί ανησυχεί ο κόσμο. Έχουμε τρόπους να γίνει αυτή η ανησυχία σε ε, ατομικές και συλλογικές δεσμεύσεις έτσι ε, ώστε ε, ο κόσμος να κινητοποιηθεί, να συνειδητοποιηθεί, να ελέγξει και τελικά να ενώσει τις δυνάμεις του για να φτάσουμε σε αυτή την πράσινη συμφωνία. Ευχαριστώ για ένα λεπτό κυρία Μέτς. Αγαπητοί συνάδελφοι, Συμφωνώντας σε τέτοιες εμπορικές συμφωνίες ε, συμφέρουμε άμεσα ε, σε αύξηση και επιτάχυνση της κατανάλωσης. Ακούσαμε το αφήγημα ότι τέτοιου είδους εμπορικές συμφωνίες οδηγούν σε ανάπτυξη. Αυτό είναι ψεύδος, πολύ λίγοι εποφελούνται, ενώ αποψηλώνονται οι παγκόσμιοι φυσικοί πόροι και ε, βοηθάμε στην καταπάτηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Στην περίπτωση της συμφωνίας Μερκοσούρ, κοιτάξτε πόσο παράλογο είναι τεράστιοι όγκοι ε, κρέατος ε, διακινούνται. Το εμπόριο κανονικά θα πρέπει να αφορά αγαθά που δεν έχει ο άλλος και το αγοράζει από κάπου. Τώρα κυκλοφορούν σε όλη την Ιφίλιο διάφορες ποσότητες κρεάτων και άλλων τροφίμων ε, χωρίς κανένα λόγο. Είναι τεράστια σπατάλη πόρων. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το βόλιο κρέας που είναι και η μεγάλη ένταση στην παραγωγή του. Πώς αυτό συνάδει με την Πράσινη Συμφωνία. Θα πρέπει εμείς ε, να πηγαίνουμε προς την άλλη κατεύθυνση, όχι να ρίχνουμε ε, λάδι στη φωτιά, βενζίνη προκειμένου. Για δύο λεπτά ο κύριος Λεμπρετών, παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε η πράσινη συμφωνία την οποία κατέθεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι πολύ φιλόδοξη, διότι έχει στόχο ουδετερότητα ως προς τον άνθρακα μέχρι το 2050. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έτσι διακηρύσει την βούλησή τη να είναι υποδειγματική στην εφαρμογή των συμφωνιών των Παρισίων. Ε, είναι πολύ αξιέπαινη η πρόθεση, αλλά η πραγματικότητα είναι τελείω διαφορετικά. Από τι συμφωνίε ελευθέρων συναλλαγών που έχουμε με όλο τον κόσμο, προδίδουμε ουσιαστικά τους στόχους που βάλαμε ήδη για το περιβάλλον. Ο καλύτερος τρόπος να καταπολεμηθεί η ατμοσφαιρική ρήπανση είναι οι μικρές αποστάσεις για να περιορίζεται η κυκλοφορία των εμπορευμάτων σε μεγάλες αποστάσεις που χρειάζεται μαζική χρήση βαρέως καυσίμου, βαρέως πετρελαίου και κυροζίνης. Το αντίθετο κάνουν ακριβώς οι συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών. Και τώρα με τη Μερκοσούρ είναι εμβληματική η συμφωνία αυτή. Το ομολόγησε και ο ίδιος ο Ιούνκερ. Είναι η μεγαλύτερη εμπορική συμφωνία που συνήψε ποτέ η Ευρωπαϊκή Ένωση πάνω από 770 εκατομμύρια καταναλωτές και 18 δισεκατομμύρια ΕΠ. Φυσικά είναι η μεγαλύτερη συμφωνία και είναι πολύ σοβαρό για το περιβάλλον γιατί η Λατινική Αμερική είναι γεωγραφικά πολύ μακριά από την Ευρώπη και θα ρηπαίνουν πάρα πολύ αυτές οι εμπορικές συναλλαγές. Στη συνέχεια, το περιεχόμενο αυτών των συμφωνιών ε, θυσιάζει πάντα την προστασία του περιβάλλοντος ε, στην ε, αγωνία που έχουμε πάση θυσία να εξάγουμε τη βιομηχανική μα παραγωγή. Και δεν είναι εξαίρεση αυτή η συμφωνία με το Μερκοσούρ. Καλά, μπορεί να υπάρχει ένα κεφάλαιο που ε, υποτίθεται ότι προάγει την ε, προστασία των δασών και τη βιωσιμότητα. Αλλά ουσιαστικά καταστρέφει περισσότερο από ποτέ τα δάση του Αμαζονίου. Καταλαβαίνετε τι εγγύηση είναι αυτή. Ε, άκρατος φιλελευθερισμός και σε αυτό το βωμό η Ευρωπαϊκή Ένωση ηθελημένα θυσιάζει στα λόμπι της αυτοκινητοβιομηχανίας, τη χημία, τη φαρμακοβιομηχανίας, των μεταφορών, των ε, επικοινωνιών και των οικονομικών υπηρεσιών το κλίμα. Και έρχεται για άλλη μια φορά να εξαπατήσει του Ευρωπαίους κηρύσσοντα άλλα στην Πράσινη Συμφωνία. Ευχαριστώ για ένα λεπτό κύριο κύριος Προκατσίνη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η σημερινή συζήτηση είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα, διότι μα δείχνει δύο διαφορετικέ όψει, δύο διαφορετικά πρόσωπα μάλλον. Πρώτα απ' όλα έχουμε την παραβολαντική σκοπιά όσων ε, έχουν κομμουνιστική ιδεολογία αλλά προσπαθούν να ξεφύγουν από αυτή και να δώσουν ένα νέο νόημα στην πολιτική τους δράση. Τελικά καταλήγουμε να βλάψουμε την οικονομία και τους εργαζομένους που μέχρι χθε λέγατε ότι θέλετε να προασπιστείτε. Ε, το άλλο πρόσωπο είναι αυτόν όσον αρχίζει να βγάζει από το στόμα του μεγάλες ηχηρές φράσεις όπως η νέα πράσινη συμφωνία, αλλά μετά σκασίλα του για την προστασία του περιβάλλοντος. Διότι ο το μόνο πράσινο που φαίνεται να ενδιαφέρει είναι το χρήμα των χαρτονομισμάτων. Και αναφέρομαι στα ευρωπαϊκά κράτη που χάρη στην ε, συμφωνία με τη Μερκοσούρ θα μπορούν πιο εύκολα να πουλάνε ε, αυτοκίνητα μεγάλου κυβισμού ε, εις βάρος των ευρωπαϊκών εταιριών που θα πληγούν ιδιαίτερα. Και βλέπουμε ταυτόχρονα τα δύο πρόσωπα να εκφράζονται εδώ όπως ένα πίνακα του Παύλου Πικάσο και αναδεικνύεται ε, ανάγλυφα η υποκρισία μας. Ευχαριστώ πολύ. Η Επόμενη ομιλήτρια για ένα λεπτό, η κυρία Σύρα Ρέγκο. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Την περασμένη εβδομάδα, εδώ στο Κοινοβούλιο, καταθέσατε την πρότασή σας για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Εκεί είδαμε πολλά ερωτηματικά και ε, πολλά αντιφατικά. Ένα βασικό θέμα είναι συμφωνίε ελευθέρων συναλλαγών, σαν αυτή που θέλετε να κυρώσετε τώρα με τη Μερκοσούρ και σημαδεύει την εμπορική μα πολιτική. Είναι πολλέ οι κριτικέ, ε, οι βάσιμε που εκφράζουν συνδικαλιστέ, αγροτοσυνδικαλιστέ, ακτιβιστέ ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ευρώπη και Λατινική Αμερική. Μεταξύ άλλων, διακινεί 88 ε, δις ε, αξίας εμπορεύματα με τις αντίστοιχες εκπομπές. Ε, παράγεται βόλιο κρέας καταστρέφοντας τον Αμαζόνιο και τα δάση. Με φυτοφάρμακα παράγονται φυτικά τρόφιμα. Και φυσικά ε, δίνεται ευλογία στις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από πλευράς του φασίστα Μπολσονάρο. Εμείς θέλουμε βιωσιμότητα και μείωση εκπομπών λέτε ότι η Ευρωπαϊκή Πράσινα Συμφωνία είναι για να μην μείνει κανένας πίσω. Να μην μείνει καμιά μεγάλη υποεθνική, πολυεθνική πίσω. Αυτό θέλετε ουσιαστικά. Ευχαριστώ. Επόμενος ομιλητής για 1,5 λεπτό, ο κύριος Κρίς Πέτερς, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία της περασμένης εβδομάδας έχουμε την πιο φιλόδοξη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, που είναι υπέρ της βιώσιμης ανάπτυξης του βιώσιμου κόσμου για τα παιδιά μας. Ε, και εκεί θα πρέπει να προβληματιστούμε και για τις οικολογικές συνέπειες της εμπορικής μας πολιτικής. Και εδώ θα πρέπει να σπάσουν κάποια ταμπού. Η γεωργία είναι ένα τέτοιο ταμπού που είναι ο ακρογωνιαίος λίθος μας για την περιβαλλοντική πολιτική και σωστά το λέμε. Αλλά οι Ευρωπαίοι αγρότες έχουν και τα πιο υψηλά περιβαλλοντικά πρότυπα παγκοσμίω. Το βόλιο κρέας που εισάγουμε ρηπαίνει περισσότερο για την παραγωγή του από ότι τον τόπιο. Αλλά και στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ρηγμένοι οι Ευρωπαίοι αγρότες. Και τολμώ να αναρωτηθώ για ποιο λόγο έχουμε δικαιώματα εισαγωγών για βόηο κρέας. 99.000 τόνοι με πολύ υψηλότερο ε, αποτύπωμα οικολογικό ε, για την παραγωγή του ε, σε σχέση με τη βελγική φυλή. Έτσι θα πρέπει να τους ε, υποστηρίζουμε με επιδοτήσεις ή μήπως να σκεφτούμε περισσότερο ένα πιο οικολογικό εμπόριο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Επόμενος ομιλητής για ένα λεπτό και μισό, ο κύριος Σάβη Λόπεθ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Σήμερα συζητούμε για μια συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Μερκοσούρ που απαιτεί συζήτηση και αξίζει συζήτηση σε βάθος και έλεγχο και θα το κάνουμε τα επόμενα χρόνια εδώ στο Κοινοβούλιο. Σημαίνει ευκαιρία για πραγματική ε, διαπεριφερειακή συμμαχία Λατινικής Αμερικής Ευρώπης. Θέλω να θυμίσω ότι αυτό θα επέτρεπε ε, να συνδεθεί το 85% ε, του πληθυσμού της Λατινικής Αμερικής με τη μεγαλύτερη αγορά στον κόσμο, που είναι η ευρωπαϊκή αγορά. Και το λέω τώρα, επειδή αλλάζει ο κόσμος και εμείς αναζητούμε συμμάχους για την προστασία της δίκαιης παγκοσμιοποίησης, χωρίς αποκλεισμούς, με την πολυμερή συνεργασία. Στη Λατινική Αμερική έχουμε ένα τέτοιο εταίρο και αξίζει τον κόπο. Ε, αυτή η συμφωνία και οποιαδήποτε άλλη ε, να χρησιμεύσει όχι για να εξάγουμε προϊόντα, αλλά για να εξάγουμε πρότυπα και κανόνες. Και ακριβώς οι εμπορικές συμφωνίες ε, για αυτό το λόγο υπάρχουν και αυτό το σκοπό εξυπηρετούν. Τώρα συζητάμε τι συμβαίνει στη Βραζιλία και ο Μπολσονάρο που βασικά εμένα μου μόνο αποτροπιασμό μου προκαλεί και συμφωνώ με αυτά που λέτε. Ε, αλλά θα πρέπει να θυμηθούμε ότι 20 χρόνια διαπραγματευόμαστε αυτή τη συμφωνία. Και υπήρξαν και άλλοι Βραζιλιάνοι πρόεδροι που διαπραγματεύτηκαν αυτή τη συμφωνία. Και τι θα κάνουμε. Η εμπορική συμφωνία τι σημαίνει. Απαιτητικού κανόνε και σταθερό πλαίσιο για να καταπολεμήσουμε την κλιματική αλλαγή και να προστατεύσουμε τη βιοπικιλότητα, ιδίω όταν πρόκειται για τον πνεύμονα του πλανήτη. Αυτό δεν θα το κάνουμε μόνοι μα. Να συμφωνήσουμε, ε, να απαιτήσουμε και να εξάγουμε όχι προϊόντα, κανόνε και πρότυπα. Γι' αυτό το σκοπό έχουμε και αυτό το σκοπό εξυπηρετούν αυτέ τι συμφωνίε. Ευχαριστώ. Για ένα λεπτό η κυρία Ρή, παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Δεν νομίζω ότι στην ουσία η συμφωνία με το η αντιβαίνει στις φιλοδοξίες μας. Ε, νομίζω αντιθέτως ότι Υπάρχουν απλώς κάποιες μικρές λεπτομέρειες ε, μέχρι να μπορέσει να δώσει πράσινο φως στο Κοινοβούλιο και ο συνάδελφος Μαντλάκεν είπε ε, και υπογράμμισε ότι χρειαζόμαστε κάτι τέτοιο. Δύο σημεία θα αναφέρω. Οι δικοί μας ε, γεωργοί πρέπει να προστατεύονται καλύτερα και γενικότερα το γεωργικό μας μοντέλο πρέπει να προστατεύεται. Ειδικά το βόλιο, η ζάχαρη που έχουν ήδη τιμές στα βάραθρα. Έχουμε την ε, Βραζιλία του Μπολσονάρο η οποία οδηγεί σε αποψήλωση την Αμαζονία. Αυτή τη στιγμή ε, ήταν ε, αυτή που απορροφούσε όλες τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Χωρίς αυτή είμαστε στο μηδέν. Οπότε πρακτικά τι κάνουμε, τι λέμε για τη συμφωνία του Παρισιού. Είδαμε τι γίνεται, έγινε στη Μαδρίτη. Δεν είναι πια δυνατόν να ακολουθούμε το business as usual. Ευχαριστώ. Ο συνάδελφος Χόισλινγκ έχει το λόγο για ένα λεπτό. Αν θέλουμε μια πράσινη συμφωνία, δεν μπορούμε να κλείσουμε αυτή τη συμφωνία. Δεν γίνεται. Την τελευταία εκατονταετία είδαμε ακριβώ ότι δεν έχουμε πια χρόνο. Έχουμε μια συμφωνία για βόλιο έναντι ε, μηχανημάτων ε, και υπηρεσιών και αυτοκινήτων. Νομίζω όμως ότι είναι η στιγμή να ξεκινήσουμε νέες ε, διαπραγματεύσεις. Έχουμε τη βιωσιμότητα και την προστασία του περιβάλλοντος. Αυτά είναι τα κεφάλαια που πρέπει να προωθήσουμε τις κυρώσεις. Ξέρουμε ότι ο Μπολσονάρο είναι ένας ε, ε, άνθρωπος ο οποίος θέλει να περάσει το φασισμό του με αυτή τη συμφωνία. Νομίζω λοιπόν ότι ε, δεν πρέπει να τον κάνουμε ήρωα μέσα από αυτή τη ε, συμφωνία και να βάλουμε στην άκρη τη συμφωνία του Παρισιού και να τα ε, διαλύσουμε όλα. Νομίζω λοιπόν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση που προασπίζεται τα ανθρωπίνα δικαιώματα πρέπει να τα πάρει όλα αυτά σοβαρά. Υπάρχουν στάνταρ και δεν μπορούμε να έχουμε τα ίδια στάνταρ. Όταν βλέπουμε τι κάνουν οι δικοί μας γεωργοί και ταυτόχρονα εισάγουμε από μια χώρα όπου τα περιβαλλοντικά στάνταρ δεν έχουν καμία σχέση σχέση όπου υπάρχουν ε, τα λοιπάσματα που απαγορεύονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό δεν γίνεται. Ευχαριστούμε ένα λεπτό, ID Bye. Ε, εδώ ο τίτλο τη συζήτηση είναι εάν τα δόγματα τη Ευρωπαϊκή Ένωση συνάδουν με το περιβάλλον που θέλουμε να προσπιστούμε. Προφανώ και όχι, διότι αυτό είναι το μεγάλο παράδοξο τη ασυνέπεια τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, θέλουμε να επιβάλλουμε στην γεωργία και την κτηνοτροφία μα ε, κανόνε όλο και πιο δύσκολου και πιο περίπλοκου και αυστηρού και που κοστίζουν. Και μετά θέλουμε όλο και περισσότερο, και πιο γρήγορα στη λογική των ελεύθερων συλλαγίων, τη Ελληνική Ένωση, τη καταργήση των δασμών και ε, τη απελευθέρωση του εμπορίου. Πραγματικά είμαστε αφελεί και ε, είναι παράδοξο αυτό που απαιτούμε. Δηλαδή, νομίζουμε ότι οι άλλε δυνάμει του κόσμου θα ακολουθήσουν τα πρότυπά μα και τι δικέ μα τι ε, επιταγέ. Όχι, δεν είναι έτσι. Υπάρχουν περιπτώσει αθέμη ανταγωνισμού. Όλο ένα και αυστηρότεροι κανόνε που πλήττουν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και των ε, γεωργών και εκτενοτρόφων μα, που δεν του προστατεύουμε. Αντί να του προστατεύσουμε, του θανατώνουμε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν πάντα το καλύτερο μαθητή στην οικολογία. Με, λιγότερο, με μείωση 16% των εκπομπών νερού του θερμοκηπίου τα τελευταία 10 χρόνια, ενώ η Κίνα έχει πάνω από και ε, αύξηση και κατα... κατηγορεί του δυτικού. Εδώ λοιπόν πρέπει να πάψουμε την υποκρισία και να προστατεύσουμε το περιβάλλον και του δικού μα παραγωγού καθώ και την οικονομία μα. Ευχαριστούμε. Παρακαλούμε αν μπορείτε. Μην μιλάτε τόσο γρήγορα στο λίγο χρόνο που έχετε πάρει από την ομάδα σας, διότι οι διερμηνείς δυσκολεύονται. Επόμενος, επόμενη, η συνάδελφος Στέκρουτ, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η συμφωνία με το Μερκοσούρ είναι σίγουρα σημαντική, όμως σήμερα μιλάμε και για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, τις επενδύσεις, την ομοθεσία, ακόμα και την ίδια τη συμπεριφορά. Το σύνθημα είναι ότι η Ευρώπη πρέπει να είναι η πρώτη ήπειρος που θα είναι ουδέτερη σε επίπεδο εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα στον κόσμο. Εντάξει, αυτό δεν θα ήταν πρόβλημα αν μιλούσαμε όμως και για τις συνέπειες, πρέπει να μιλάμε με γεγονότα, να μιλάμε για τα υπέρ αλλά και για τα κατά. Αυτή η μεταμόρφωση θα έχει μεγάλο κόστος, ενεργειακό κόστος, ε, το οποίο επίσης θα μειώσει την ανταγωνιστικότητά μας. Και με ένα τέτοιο εγχείρημα θα μπει και ένας ε, ε, συνοριακός ε, φόρος για τα καύσιμα. Υπάρχουν εμπορικές διαφιλονικίες στον κόσμο. Εμείς λοιπόν ρισκάρουμε να μειώσουμε την ευημερία μας και τον τρόπο ζωής μας. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό για μας να υπογραμμίσουμε ότι δεν είναι το εμπόριο που τα ρυθμίζει όλα. Αυτό που τα ρυθμίζει όλα θα ήταν η πυρηνική ενέργεια και ε, τα αντίστοιχα θέματα. Ο κύριος Ουάλλας ε, για ένα λεπτό. Ε, πρόεδρε, κύριε Χόγκαν, αυτή η συμφωνία βάζει σε προτεραιότητα το κέρδος για τους επενδυτές και τις εταιρείες, ενώ μειώνει τα στάνταρ για τους εργαζόμενους, τους γεωργούς και τους πολίτες. Ειδικά οι Ευρωπαίοι γεωργοί θα πρέπει να ανταγωνιστούν με εισαγωγές από τεράστιες επιχειρήσεις στην Μερκοσούρ που χρησιμοποιούν φυτοφάρμακα, αντιβιωτικά και ορμόνες που απαγορεύονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Πράσινη Συμφωνία λέει ότι η γεωργία μας είναι το κλειδί στη μετάβαση. Η ε, στρατηγική Farm to Fork στην ουσία μας ε, οδηγεί στο να προσπαθήσουμε για τη βιοπικιλότητα, να διασφαλίσουμε μια αξιοπρεπή ζωή για τους αγρότες και τις οικογένειές τους. Για όνομα του Θεού, τι έχει να κάνει η Συμφωνία Μερκοσούρου με αυτό. Ε, έχουμε μια λανθασμένη διπλωματία όταν οι Αργεντινοί ε, ε, έχουν μπλοκάρει και άλλες τέτοιες χώρες έχουν μπλοκάρει το COP25 Λέμε ότι οι μη βιώσιμες δραστηριότητες δεν πρέπει να συνεχίσουν, όμως ο, πρόεδρος, ο Υπουργός Περιβάλλοντος της Βραζιλίας στην Μαδρίτη είπε ότι ούτε ένα Τέτρο δεν έχει κοπεί στην Αμαζονία. Το πιστεύετε αυτό που λέει. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Σμιτ Πάουα, για 1,5 λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Μια μοντέρνα σύγχρονη γεωργία βιώσιμη χρειάζεται βοήθεια ε, ε, για τις οικογενειακές επιχειρήσεις και αυτό θα πρέπει να λέει η Πράσινη Συμφωνία για τις συμφωνίες ελευθερών συναλλαγών. Αυτή η διπλωματία της Πράσινης Συμφωνίας θα εφαρμοστεί και στους εμπορικούς εταίρους και αυτό πώς θα το εγγυηθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι δεν θα έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά. Πού θα χαράξετε κόκκινες γραμμές θα πρέπει να έχουν και οι άλλες χώρες τόσο υψηλά πρότυπα περιβαλλοντικά, αν είμαστε σοβαροί με τη συμφωνία αυτή την πράσινη. Ε, ε, και επιτρέψτε μου να αλφιβάλλουμε γι' αυτό, για την ε, παραγωγή και τη βιώσιμη παραγωγή εκεί. Δεν έχουμε τους ίδιους κανόνες. Ποια στρατηγική έχουμε για τις πρωτεΐνες θα την ε, καθιερώσουμε αυτή στην Πράσινη Συμφωνία. Βλέπε εισαγωγή σόγιας. Θα πρέπει τα τρόφιμα και οι ζωοτροφές να πηγαίνουν έρχονται πάνω από τον Ατλαντικό. Και ε, θα βάλουμε σήμανση ε, στα τρόφιμα για να ξέρει ο καταναλωτής τι αγοράζει και να αποφασίζει αν θέλει να αγοράσει ντόπιο ή εισαγόμενο. Εμάς στην Αυστρία μας ενδιαφέρει πάρα πολύ η προστασία του περιβάλλοντος. Είναι η ίδια μας η ζωή. Ε, και κάνουμε πολλή δουλειά. Εγώ είμαι από την Αυστρία αγρότης, αγαπητέ κύριε Επίτροπε. Ε, χρειαζόμαστε όμως σταθερότητα, ένα συγκεκριμένο πλαίσιο ε, και να πιάνουν τόπο οι υπηρεσίες που προσφέρουμε στο γενικό σύνολο. Θα πρέπει να αμοιβόμαστε γι' αυτό και στο κάτω-κάτω πρόκειται για την ίδια την επιβίωση μιας ολόκληρης επαγγελματικής ομάδας. Ο κύριος Ντάντι για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Επίτροπε, πραγματικά μένω άναυδο, διότι σήμερα η πράσινη πρότεινα να γίνει συζήτηση όχι γενική, θεματική για τι ευθύνε τη Ευρώπη και τη σχέση τη πράσινη συμφωνία με τι εμπορικέ, αλλά ειδικά για το Μορκοσούρ. Πρώτα απ' όλα, μερικά δεδομένα. Πρώτα απ' όλα, η Ευρώπη είναι το 90% του συνόλου των ε, ρήπων. Ε, ενώ ε, οι πέντε χώρε τη Μερκοσούρ είναι, έχουν πολύ μεγαλύτερα ποσοστά για τα εκπομπή του θερμοκηπίου. και μάλιστα με πολύ χαμηλή πυκνότητα πληθυσμού και πολύ μεγάλε ε, δασόδει περιοχέ. Επίση, το κεφάλαιο βιώσιμη ανάπτυξη που είναι καθοριστικό στη Συμφωνία Μερκοσούρ. Είναι μια εγγύηση για την προστασία τη βιοπικιλότητα, για την προστασία από την αποψήλωση και για την τήρηση των υποσχέσεων που έχουν δώσει οι κυβερνήσει αυτέ με την Συμφωνία και τη Διάσκεψη των Παρισίων ε, την COP24. Εδώ λοιπόν πρέπει να δούμε τις ε, ε πολιτικές ε, υποβάθμισης τι άθλιε πολιτικέ του Πρόεδρου Μπολσονάρου, ε, οι οποίε δεν μπορούν να συνεχίσουν, όμω σε κάθε περίπτωση η στάση των Πρασίνων κρίνω ότι είναι τελείω ασυνεπή. Ευχαριστούμε. Επόμενο, ο κύριος Κέλεχερ, για ένα λεπτό. Σας καλωσορίζω, καλωσορίσω, κύριε Χόγκαν, στην ε, ναι, σας θητεία θα είναι μια προσ πρόκληση για σας μέσα σε αυτό το πλαίσιο της πρόθεσης της παγκόσμιας οικολογίας. Έχουμε μία ατζέντα για το κλίμα, αλλά πρέπει όχι μόνο εδώ να την έχουμε, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. Την ίδια στιγμή θα ρίνουμε μία εμπορική συμφωνία με την Βραζιλία, την ε, Ουρουγουάη, την Παραγουάη και την Αργεντινή, η οποία ε, στην ουσία βάζει στην άκρη το γεγονός ότι τόσα δάση στην Αμαζονία χάνονται, ότι εξαφανίζεται η βιοπικιλότητα και στέλνει το μήνυμα στον κόσμο ότι η Ευρώπη δεν είναι τόσο σοβαρή όσο θα έπρεπε για την κλιματική αλλαγή. Την περασμένη εβδομάδα ε, αποφασίσαμε κάποια πράγματα και την ίδια στιγμή υποσκάπτουμε τη θέση μας ε, γιατί ε, μιλάμε για μια συμφωνία η οποία υποσκάπτει όλα όσα υπάρχουν στην πράσινη ατζέντα. Πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι και ειλικρινεί. Αυτή εδώ η συμφωνία υποσκάπτει τις βασικές αρχές ε, που προωθούμε εμείς στην Ευρώπη σε επίπεδο περιβάλλοντος και δεύτερον και πολύ σημαντικό την γεωργική μας βιομηχανία. Ευχαριστώ. Ο συνάδελφος Χόλμγκρεν έχει το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εχθές ε, στη Σουηδία η κυβέρνηση, χάρη στο Πράσινο Κόμμα της Σουηδίας, αποφάσισε σε όλους τους πολιτικούς ε, τομείς να τεθεί ένα στόχο σε σχέση με το κλίμα. Αυτό θα έπρεπε να είναι προφανές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ειδικά μέσα στα πλαίσια των εμπορικών συμφωνιών που είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να επηρεάσουμε την κλιματική πολιτική που ε, διάγουν οι άλλες χώρες. Αυτός είναι ο τρόπος, ίσως ο μοναδικός τρόπος για να έχουμε επιρροή στις τρίτες χώρες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα έπρεπε ίσως να έχει ποτέ σχέσεις εμπορικές με χώρες που δεν υποστηρίζουν τη Συμφωνία των Παρισίων και που δεν δουλεύουν προς την πραγμάτωσή της. Ε, νομίζω ότι εδώ εμείς ως ομάδα θα πρέπει να είμαστε <clears throat> οι πιονέροι στο θέμα της κλιματικής αλλαγής. Πρέπει να δράσουμε σε όλα τα επίπεδα ε, και σε αυτή τη θητεία, σε αυτά τα πέντε χρόνια πρέπει να δράσουμε γιατί ο κίνδυνος ε, είναι να είναι η τελευταία μας θητεία. Ευχαριστώ, συνάδελφος Ρος, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συνάδελφε, Επίτροπε, την περασμένη εβδομάδα ο κύριος Τίμερμανς παρουσίασε την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία του. Εκεί έχει μια στρατηγική κατά της κτηνοτροφίας. Ε, έχουμε ε, στην Ευρώπη απαγορεύσει διάφορα φυτοφάρμακα και ε, την κτηνοτροφία σε κλωβοστοιχίες. Αλλού όμως δεν ισχύουν αυτοί οι κανόνες και με τη συμφωνία Mercosur τώρα θα έχουμε τρόφιμα στο πιάτο μας από χώρες όπου δεν ισχύουν αυτοί οι κανόνες. Αυτά είναι τελείως αντιφατικά πράγματα. Η συμφωνία με τη Mercosur είναι μια στρατηγική που λέει σας δίνουμε αυτοκίνητα, μας δίνετε γελάδια. Τη Βόλιο Κρέας δεν βγαίνει αυτή η εξίσωση. Ταυτόχρονα όλοι οι αγρότες στα κράτη-μέλη και στη δική μου χώρα, την Ολλανδία, πλήττονται από τον αθέμητο ανταγωνισμό. Και φυσικά πληρώνει την ύφη και ο καταναλωτής. Ε, θα πρέπει ε, να αναθεωρήσουμε αυτή την ε, πολιτική με τις τόσες αντιφάσεις. Ευχαριστώ για Ρούμπας για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε, κυρία Κύριε Επιτροπέ, σήμερα αντιμετωπίζουμε ένα τεράστιο δίλημα. Εκτιμάται ότι η συμφωνία με τις χώρες Μερκοσούρ θα μας δώσει 90 19 ε, ευρώ παραπάνω στο ΑΕΠ μας 19 δις ευρώ παραπάνω, 8 δις ευρώ παραπάνω στις συναλλαγές ε, αγαθών και προϊόντων και ακόμη περισσότερο με τις υπηρεσίες. Αυτό επίσης μπορεί να οδηγήσει σε περισσότερη αποψήλωση της περιοχής του πλανήτη μας, του, του Αμαζονίου, των δασών του Αμαζονίου, προκειμένου να γίνει περισσότερος χώρος για την καλλιέργεια σόγιας. Ε, έχουμε λοιπόν την πρόταση αυτή να χρησιμοποιήσουμε τη συγκεκριμένη συμφωνία για να ασκήσουμε πίεση και να ζητήσουμε από τις χώρες Μαρκοσούρ να αλλάξουν τη στάση τους και την πολιτική τους. Αυτό όμως μπορεί να συμβάλλει ταυτόχρονα σε περισσότερες εκπομπές ε, αέριων του θερμοκηπίου λόγω των μεταφορών. Πραγματικά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη συμφωνία αυτή για να πιέσουμε τους εταίρους μας, τους συνομιλητές μας, να συμμορφωθούμε τα δικά μας πρότυπα ως προς τα φυτοφάρμακα, την ευζοία των ζώων, την ασφάλεια των τροφίμων μας, διότι όλα αυτά τα πρότυπα οφείλουν να τα τηρούν οι Ευρωπαίοι γεωργοί και ακτινοτρόφοι. Μιλάμε για μια μορφή ε, πίεση που πρέπει να του ασκήσουμε σίγουρα, αλλά δεν είναι η μόνη. Από την άλλη έχουμε και τι τράπεζε, τις τράπεζες που επενδύουν ε, από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού ε, με διαφορετικά πρότυπα Ποιο ε, θα πρέπει να είναι λοιπόν ε, το βασικό ε, διακύβευμα της Πράσινης Συμφωνίας εδώ θα υπάρχει και μια περίοδος μετάβασης που θα μας επιτρέψει να δούμε αν τηρούνται τα πρότυπα. Μάλιστα, ευχαριστούμε. Επόμενος ομιλητής ο κ. Ζήντλ για ένα λεπτό. Κυρία Πρόεδρε, μια εμπορική συμφωνία με το Μερκοσούρ ε, στην ουσία θα ανοίξει την Λατινική Αμερική για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η παραγωγή από την Βραζιλία που μπορούν με χαμηλό κόστος να παράγουν μεγάλες ε, ποσότητες μπορούν να προωθήσουν τις εξαγωγές τους, να αυξήσουν την παραγωγή τους και αυτό να έχει μεγάλες συνέπειες ε, για το περιβάλλον και την εσωτερική αγορά τη Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βλέπουμε τη χρήση των ε, φυτοφαρμάκων στη Μερκοσούρο ως ένα γνωστό πρόβλημα, πράγματα που είναι απογορευμένα στην Ευρώπη. Υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα στάνταρτς ε, τα οποία δεν τηρούνται στα προϊόντα της Λατινικής Αμερικής. Επίσης, οι πρακτικές πυρκαγιών για την δημιουργία καλλιεργήσιμων εκτάσεων είναι καταδικαστές πρέπει λοιπόν ε, αυτό έχει πετύχει η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα από αυτό ε, τη συμφωνία να μην τα θάψουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ο συνάδελφος Φόντεν έχει το λόγο για ένα... Η συνάδελφο Φόντεν έχει το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Αυτό το κοινοβούλιο ε, δέχτηκε μια υπόσχεση για μια ριζοσπαστική πράσινη συμφωνία. Υπάρχουν οι νέοι που κοιτούν προς εμάς γιατί πήραν αυτή την υπόσχεση. Αν όμως αυτό σημαίνει τουλάχιστον κάτι, αυτή η συμφωνία θα πρέπει να καλύπτει όλες τις πτυχές της νομοθεσίας. Οποιαδήποτε συμφωνία διαπραγματευόμαστε, όχι απλώς τη Μερκοσούρ. Η μόχλευσή μα θα είναι μεγαλύτερη ε, πριν υπογράψουμε. Πρέπει οι στόχοι για το περιβάλλον να είναι πολύ, καλή, πολύ πιο ψηλά από ότι το βόλιο κρέα στα ράφια του σούπερ μάρκετ. Οι νέες εμπορικέ συμφωνίε πρέπει να εγγυώνται την εφαρμογή αυστηρή περιβαλλοντική νομοθεσία, ε, τη δημοκρατία και τα δικαιώματα των πολιών. Η συμφωνία για τη Μερκοσούρ ήταν η καλύτερη ευκαιρία που είχαμε ποτέ για να κερδίσουμε εγγυήσει για την προστασία του Αμαζονίου. Αν ε, εννοούμε αυτά που λέμε και ότι θέλουμε να βάλουμε προτεραιότητα το κλίμα, ήρθε η ώρα να κάνουμε πράξη αυτά που λέμε. Χρειάζεται χρόνος για να διαπραγματευτούμε μια συμφωνία. Στο μεταξύ με τις διαπραγματεύσεις αυτές το κλίμα έγινε επίγουσα κατάσταση και πρέπει να είναι η προτεραιότητά μας. Ευχαριστώ. Ένα λεπτό. Συνάλφος Βίνερ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, Επίτροπε, ε, εάν ακούσατε όσα υπόθηκαν εδώ, θα πρέπει να καταλάβετε ότι η Ευρώπη δεν πρέπει καμία, να συνάψει καμία συμφωνία με, τη Μερκοσούρ, με τις χώρες Μερκοσούρ. Πρώτα απ' όλα γιατί έχουμε ηθική υποχρέωση να ακούσουμε τις φωνές από την Ευρώπη και να σκεφτούμε ότι αυτή η συμφωνία με τη Μερκοσούρ είναι σαφής Διαβάστε τη λέγεται σήμερα. Δεν υπάρχει καμία συμβατότητα με την πράσινη συμφωνία τη Ευρώπη και τη συμφωνία Μερκοσούρ. Και είναι πολλοί οι λόγοι. Η προστασία του περιβάλλοντο από το κλίμα, η προστασία των μικρών κτηνοτρόφων και γεωργών, ε, η βιοπικιλότητα, η αποψήλωση του Αμαζονίου, η παραγωγή τροφίμων με τεράστια παραγωγική μηχανή. Εδώ λοιπόν η ανθρωποί αλλά και οι μικροί γεωργοί και ε, δεν θα υποστηριχθούν από αυτή τη συμφωνία, μόνο τα μεγάλα αγροκτήματα. Ευχαριστούμε. Επόμενος ε, η κυρία Κολά Οστερλέ για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, συνάδελφοι, οι εμπορικέ μα συναλλαγέ και οι εισαγωγέ μα θα πρέπει να μην είναι τροχοπέδι για την συλλογική μα μάχη κατά των κλιματικών αλλαγών. Η συμφωνία με τι χώρε Μερκοσούρ είναι όμω μια οπισθοδρόμηση, διότι θα καταργήσει του δασμού για 82%, 92% των προϊόντων από τη Μερκοσούρ που ε, εισάγονται προ την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εδώ τίθεται θέμα ισότητα και ισοτιμία. Για να φτάσουμε την ουδετερότητα προ τι εκπομπέ ε, διοξιδίου του άνθρακα το 2050. Θα πρέπει οι ευρωπαϊκέ εταιρείε να αναλάβουν επιπλέον υποχρεώσει για τη μείωση των ε, κομπών νερού του θερμοκηπίου. Δεν μπορούμε να τι τιμωρούμε ε, επιτρέποντα εισαγωγέ που δεν θα έχουν να ακολουθήσουν τέτοια πρότυπα. Οι μηχανισμοί μετάβαση, ο άνθρακα με τα σύνορα και όπω προβλέπει η Πράσινη Συμφωνία πρέπει να προβλεφθεί αμέσω με απλού εύληπτου κανόνε ε, και μια απλή πορεία που θα πρέπει όλοι να μπορούν να ακολουθήσουν. Πρέπει να απορρίψουμε κάθε θέμα τον ανταγωνισμό. Πώ θα επιβάλλουμε ακόμα περισσότερου κανόνε στου και γεωργού μα και θα ανοίξουμε τι πόρτε σε γεωργική παραγωγή που δεν σέβεται κανένα κανόνα. Οι Ευρωπαίοι καταναλωτέ, οι υγειονομικοί μα κανόνε είναι πράγματα που θα σεβαστούμε, είναι θέμα δημόσια υγεία. Και πρέπει να σκεφτούμε την ε, μηχανή παραγωγή μα και του ε, παραγωγού μα με ίσου κανόνε στο παγκόσμιο προσκήνιο. Επίση, θέλουμε μια βιώσιμη διαχείριση των πόρων μα. Πρέπει να προβλέψουμε ρήτρε δεσμευτικέ για τι εμπορικέ μα συμφωνίε που να σέβονται όσα προβλέπει η Συμφωνία των Παρισίων για την προστασία του, από, το, από τι κλιματικέ αλλαγέ και για την προστασία των δασών. Πρέπει να πάψει η αποψήλωση στα τροπικά δάση του Αμαζονίου. Δεν μπορούμε να δεχτούμε μια συμφωνία που δεν ε, ε, συναντεί με τι υποσχέσει και τι δεσμεύσει που ανέλαβε η πρόεδρο ε, Ursula von der για όσα θέλουν να ισχύσει στην εσωτερική μα αγορά. Ευχαριστούμε κυρία Ρενά για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μα παρουσίασε τι φιλοδοξίε τη για τα κλιματικά ζητήματα με την Πράσινη Συμφωνία και χαίρομαι γι' αυτό. Όμω, πώ γίνεται ταυτόχρονα η ίδια Επιτροπή να δικαιολογήσει την υπογραφή μια τέτοια συμφωνία όπω αυτή που έχουμε μπροστά μα, μια συμφωνία που είναι παλιά γενιά, την οποία είχαμε αντιπραγματευτεί πριν από 20 χρόνια και σαν να μην συμβαίνει πλέον τίποτα. Πού είναι η πολιτική μα συνοχή όταν αυτή η συμφωνία και για το κλίμα και για την αποψήλωση και για του ηθιγενεί πληθυσμού και για την επικοινότητα και τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν κάνει τίποτα. Δεν προσπα... πρέπει να προσπαθείτε να μα πείσετε ότι το κεφάλαιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη ανάπτυξη είναι εγγύηση για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Δεν ισχύει αυτό και το γνωρίζετε. Να είμαστε συνεπεί με του εαυτού μα. Να είμαστε συνεκτικοί ε, και ειλικρινεί. Γιατί το κεφάλαιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη εξαιρείται από του μηχανισμού διευθέτηση των διαφορών κράτου με κράτο. Που αυτή τη στιγμή ισχύει για όλε μα τι εμπορικέ συμφωνίε στο σύνολό του. Και όταν πρόκειται για ανθρώπινα δικαιώματα, γιατί τα ανθρώπινα, τα δικαιώματα μάλλον τη βιώσιμη ανάπτυξη, εκεί δεν υπάρχει δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί αυτό ο μηχανισμό επίλυση διαφορών. Ε, άρα, για να είμαστε συνεπεί. Σας καλώ να διαβάσετε όσα λέγονται ε, από το Νταβός ε, που λέει ότι μια εταιρεία θα πρέπει να αντιλαμβάνει την ευθύνη ε, περιβαλλοντικά και κοινωνικά. Κύριε Πίτροπε και κυρία εκπρόσωπε του Συμβουλίου, σας καλώ να είστε λιγότερο ιδεολόγοι σε ό,τι αφορά τι εμπορικέ συμφωνίες και να σέβεστε αυτά που οι ίδιε εταιρείε κάνουν σήμερα ω προ τι προ του περιβαλλοντικού μα κανόνε. Ευχαριστούμε. Επόμενο, ο συνάδελφο Πάετ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Αυτή τη στιγμή που έχουμε τις γεωπολιτικές αλλά και στους εμπορικούς πολέμους ε, και την αναδυόμενη απειλή των ε, πολυμερών σχέσεων βλέπουμε ότι η συμφωνία Μερκοσούρ δείχνει μία δέσμευση και από τις δύο πλευρές ως προς κανόνες που βασίζουν το διεθνές εμπόριο. Θα δώσουν ε, επίσης στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις τη δυνατότητα να ξεδιπλώσουν το οικονομικό δυναμικό τους ταυτόχρονα. Το θέμα του περιβάλλοντος και της κλιματικής αλλαγής χρειάζεται παγκόσμια απάντηση. Σε κάθε λοιπόν συμφωνία η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να εφαρμόζει και να ενδυναμώνει τις δεσμεύσεις της για την βιώσιμη ανάπτυξη. Η Μερκοσούρ δεν πρέπει να είναι εξαίρεση. Είμαστε στο σωστό δρόμο με την Αργεντινή, τη Βραζιλία, την Παραγουάνη και την Ουρουγουάη όταν ζητούμε ε, για την εφαρμογή της συμφωνία των Παρισίων. Ευχαριστώ. Ο συνάδελφο, η συνάδελφος ο Σάλιβαν έχει το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλώ ήρθατε, Επίτροπε Χόγκαν. Χαίρομαι που αυτή η συζήτηση γίνεται σήμερα εδώ και ξεκίνησε από την δική μου, την ομάδα των Πρασίνων. Πολλές φορές ε, δεν έχουμε καταφέρει να βελτιώσουμε τον κόσμο μέσα από την εμπορική πολιτική. Απλώς κάνουμε συμβεβασμούς μέσα από ντυλ που έχουν να κάνουν με το κέρδος ε, και τα μη βιώσιμα φθηνά προϊόντα. Δεν μπορεί η Συμφωνία Μερκοσούρ να είναι συμβατή με την Πράσινη Συμφωνία. Πώς ε, θα μπορούσε να, είναι αυτό, να γίνει αυτό αν έχουμε τόσες φθηνές εισαγωγές με καταστροφή των τροπικών δασών, να έχουμε εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων και όχι του κλίματος. Έχουμε στην ουσία ε, μία διπλή γλώσσα. Ε, μιλάμε για ε, βιώσιμη γεωργία και την ίδια στιγμή εισάγουμε προϊόντα που δεν συμφωνούμε αυτή την πρακτική. Χρειαζόμαστε να, υποχρε... να σεβαστούμε τις υποχρεώσεις από τη Συμφωνία των Παρισίων, τα δικαιώματα των εργαζομένων και τα βασικά στοιχεία της Πράσινης Συμφωνίας. Επίσης, ε, δεν θα πρέπει να δημιουργήσουμε χάος ε, στην Ευρωπαϊκή Γεωργία. Ήδη η γεωργοί μας είναι αντιμέτωποι με απαράδεκτα χαμηλές τιμές. Ευχαριστώ. Η συνάδελφος Φιρκούνεν για 1,5 λεπτό είναι η επόμενη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συζητούμε για την συμβατότητα του Μερκοσούρ με ε, την Πράσινη Συμφωνία. Κύριε Επίτροπε Χόγκαν, το θέμα δεν είναι ε, να είναι συμβατά ή ασύμβατα. Δεν είναι απλώς συμβατές οι δύο συμφωνίες, αλλά η ασυμβατα δεν ειναι απλως συμβατες σε δυο συμφωνιες αλλα η συμφωνια με τη Μερκοσούρ είναι τμήμα της πράσινης συμφωνίας. Η Ευρώπη πρέπει να απαγκιστρωθεί από το διοξίδιο του άνθρακα, αλλά αυτό θα πρέπει να είναι βιώσιμο οικονομικά, κοινωνικά, αλλά και περιβαλλοντικά. Οικονομικά και κοινωνικά ε, το είπα, χρειαζόμαστε μια Ευρώπη βιώσιμη και ένα βιώσιμο πλανήτη γενικότερα. Δεν αρκεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να καταφέρει να είναι ουδέτερη ως προς το διοξίδιο του άνθρακα μέχρι το 2050. Πρέπει να την ακολουθήσουν και άλλες χώρες. Οι δικές μας εκπομπές είναι το 10% μόνο των παγκόσμιων εκπομπών. Θα πρέπει να μας μιμηθούν και να μας ακολουθήσουν και οι άλλες περιοχές του κόσμου. Στη Μαδρίτη δυστυχώς δεν προχωρήσαμε όσο θα θέλαμε. Τώρα έχει πολύ μεγάλη σημασία η Κίνα, η Ινδία, η ΗΠΑ τα επόμενα χρόνια να μας ακολουθήσουν και να δεσμευθούν υπέρ του κλίματος, με διεθνείς συμφωνίες. Έχει πολύ μεγάλη σημασία όλα αυτά να συμπεριληφθούν στις συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών. Και η Συμφωνία Μερκοσούρ έχει ένα κεφάλαιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Θα πρέπει οπωσδήποτε να παρακολουθούμε πώς θα εφαρμόζεται αυτή η συμφωνία. Ευχαριστώ. Η συνάδελφος Καρβαλιάης, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρία Πρόεδρε, Έχουμε σχέσεις περίπλοκες, σχέσεις αλληλεξάρτησης, αλλά βλέπουμε και τάσεις με τις χώρες Μερκοσούρα, αλλά βλέπουμε και τάσεις προστατευτισμού. Οι εμπορικές μας συμφωνίες πρέπει να είναι ευκαιρία και για να αυξήσουμε τις εξαγωγές μας και για να μεγαλώσουν, να αυξηθούν οι θέσεις απασχόλησης. Πρέπει να αφήσουμε χώρο στο διάλογο και, συνεννόησης, και χώρο συνεννόησης με τον κόσμο. Πρέπει να υπερισχύσουν οι αξίες της βιώσιμης ανάπτυξης των ανθρώπινων και εργασιακών δικαιωμάτων, των των προτύπων, των ε, κανόνων και την ζωική ευζοία, τη επιστημική ασφάλεια, του δίκαιου εμπορίου. Πρέπει να έρθουμε κοντά με χώρε και γεωγραφικά με και πλάτη που πρέπει να ακολουθήσουν στόχου ακρέπενου παρόμοιου με του δικού μα. Εδώ οι πολιτικοί στόχοι που συμπεριλαμβάνονται στη συμφωνία με το Μερκοσούρ, καθώ και η αμοιβαιότητα, ε, η κοινή ευθύνη για να υλοποιηθούν τα τη συμφωνία των Παρισίων, η, ε, η το ειδικό κεφάλαιο για τα οδηγούμενα προς ε, εξάλληψη είδη χλωρίδας και πανίδας πρέπει να παραμείνει ε, όχι απλώς μια άσκηση ρητορική, αλλά να γίνει πράξη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να κοιτάξει με όλα τα εργαλεία ελέγχου που διαθέτει να ε, παρακολουθεί αυστηρά το κατά πόσον ε, πληρούνται οι κανόνες που συμφωνήθηκαν και αν υπάρχουν παραβιάσεις που δεν είναι συμβατές με την οικολογική, μας, με την οικολογική διάσταση της συμφωνίας. Ευχαριστούμε. Επόμενη η συνάδελφος Ντεπανέ Γκρουνένμπεργκ Για ένα λεπτό. Κυρία Πρόεδρε, κύριε Χόγκαν, στην οικολογική μας κρίση που βρίσκεται αυτή τη στιγμή η ανθρωπότητα, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να κοιτάξει αν θα κλείσει μια συμφωνία που έχει ειδικό στόχο να επιτρέψει ε, να εισάγεται ζώιο, βόλιο κρέας και σόγια. Επίσης, Πρέπει να μην επιτρέψουμε και άλλε γεωργικέ εκτάσει να δημιουργηθούν από την υποψήλωση των δασών του Αμαζονίου. Ο Μπολσονάριο έχει πει ότι δεν τον ενδιαφέρει η προστασία από τι κλιματικέ αλλαγέ. Τον ενδιαφέρει κάθε ευκαιρία για να γίνει και άλλο εμπόριο, ε, να υπάρξουν και άλλε επιχειρήσει. Εδώ λοιπόν διακυβεύεται η, απολυ... η ε, εξαφάνιση τη βεπικιλότητα. Ε, το τροπικό δάσο τη Αμαζόνα, του Αμαζονίου, είναι η αιστεία με... τη βεπικιλότητα όλου του πλανήτη. Με χιλιάδε είδη χλωρίδα, πανίδα, πουλιά, ζώα και φυτά. Ε, τα πιο σπάνια είδη φυτών, δέντρων και λόχμη ε, είναι στον Αμαζόνιο αυτή τη στιγμή, σε όλο τον πλανήτη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν έχει καθήκον αυτό να μην το επιτρέψει. Η συμφωνία με τη Μαρκοσούρ, όπω ε, στη μορφή που έχει σήμερα, αντιφάσκει με όλα όσα έχουμε προβλέψει για την προστασία του περιβάλλοντο. Ευχαριστούμε, κυρία Κομπούλα Νάτρη, για ένα λεπτό. Με συγχωρείτε, με συγχωρείτε μου διέφυγε. Ο κύριος Ντιντιέ. Με συγχωρείτε. Κυρία Πρόεδρε, υπάρχουν σοβαρές πολιτικές ασυνέπειες και οι ευρωπαϊκοί ε, λαοί δεν αντέχουν πλέον δεν τις υποφέρουν. Η συμφωνία με τους εταίρους μας της Βραζιλίας, της Αργεντινής, της Παραγουάης και της Ουρουγουάης είναι ακόμη μια ε, τέτοια απόδειξη. Σε μια φάση που η Ευρώπη υπόσχεται να ε, περάσει στην καινοτομία με ε, εισαγωγές από χώρες που δεν σέβονται τους ίδιους περιβαλλοντικούς κανόνες, πώς να διανοηθούμε ότι κάποιοι σε συνθήκες πλήρους αδιαφάνειας μπορούν να επιτρέψουν σε χώρες της Λατινικής Αμερικής να κατακλείσουν την ευρωπαϊκή αγορά με τρόφιμα ή με, που είναι γεμάτες από ουσίες οι οποίες απαγορεύονται στους δικούς μας γεωργούς και εκτινοτρόφους. Σε αυτό το παράλογο της γεωργίας και εκτινοτροφίας θα δημιουργηθεί και ένα κοινωνικό παράδοξο όπου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν θα πρέπει να συμβάλλει, δεν θα πρέπει να γίνει συνένοχος. Ε, το βλέπουν οι πολίτες. Πώς θέλετε να γυρίσουμε να πούμε στους κτηνοτρόφους ε, βοηδών που ήδη έχουν βρεθεί σε κατάσταση απελπισίας και κάθε χρόνο πρέπει να ασχοληθούνται να ασχολούνται και να αντιμετωπίσουν την εισαγωγή 100.000 ε, τόνων εκατοντάδων χιλιάδων μάλλον τόνων βόη από την ε, Λατινική Αμερική που είναι τίγκα στα αντιβιωτικά. Πώς να τους επιτρέψουμε να κάνουν κάτι για τα τρόφιμα που ρούνται στα σούπερ μάρκετ που είναι όλα επικίνδυνα για τα παιδιά τους, για τις οικογένειές τους. Και τι να κάνουν οι άνθρωποι αυτοί στις οικογενειακές εκμεταλλεύσεις που δίνουν ζωή ε, κάθε μέρα για να επιβιώσουν ως προς την επισητιστική ασφάλεια ε, και με αυτές τις συμφωνίες των παρασκηνίων πρέπει να απαντήσουμε με το πνεύμα ευθύνης και, και ε, λογικής που πρέπει να μας ε, ε, που πρέπει να πριτανεύσει. Δεν πρέπει να είμαστε πλέον οι αφελείς της παγκοσμιοποίησης. Πρέπει επιτέλους οι ευρωπαϊκοί λαοί να ξαναπάρουμε στα χέρια το πεπρωμένο μας. Ευχαριστώ. Τώρα έχει η κυρία Νάτρη. Κύριε Πρόεδρε, το ερώτημα είναι αν η Πράσινη Συμφωνία και η Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου Μερκοσούρ συνάδουν. Η ε, συμφωνία με τη Μερκοσούρ έχει δεσμευτικό χαρακτήρα για την εφαρμογή της Συμφωνίας των Παρισίων. Όμως αυτή η δέσμευση γίνεται μέσα στο κεφάλαιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Έτσι δεν υπόκειται σε κυρώσεις. Αν λοιπόν η συμφωνία κυρωθεί ως έχει, στην ουσία οι Βρυξέλλες ε, κάνουν πίσω ως προς τις δεσμεύσεις τους ε, για την Συμφωνία των Παρισίων. Έχουμε ε, αποψήλωση των δασών και δεν πετυχαίνουμε τους στόχους μέχρι το 2030 και δεν είμαστε πιστοί φυσικά σε αυτά που λέμε. Εμείς όπως μάθαμε την περασμένη εβδομάδα στη Μαδρίτη στο COP25 αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Όμως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δεσμευτεί ότι θα κάνει την Συμφωνία των Παρισίων ένα βασικό κομμάτι όλων των μελλοντικών εμπορικών συμφωνιών. Είναι ένα οσιώδες στοιχείο μιας ε, συμφωνίας. Αυτό θα οδηγεί σε κυρώσεις εμπορικές. Προτείνω λοιπόν να βρούμε μια λύση. Τώρα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να, να συνδέσει με όρο αυτή τη συμφωνία και να πει ότι η Συμφωνία των Παρισίων πρέπει να είναι ουσιαστικό κομμάτι της συμφωνίας με το Μερκοσούρ. Αυτή η λύση θα βοηθήσει να, μας... να προοδεύσουμε προς τον τομέα της κλιματικής αλλαγής. Ευχαριστώ. Ο συνάδελφος Πόλτσακ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Ε, αυτή η συζήτηση οδηγεί σε πολλά διέξοδα. Βλέπουμε ότι αυτή η συμφωνία μας οδηγεί σε πολλά διέξοδα. Όμως ας μείνουμε στα γεγονότα. Είναι σημαντικό οι χώρες του Μερκοσούρ και η Ευρωπαϊκή Ένωση που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία του Παρισίου να ε, προχωρήσουν ε, σωστά. Βασικά στην Βραζιλία, ε, στη Βραζιλία υπάρχει αποψήλωση των δασών. τι κάνουμε λοιπόν σε αυτό το θέμα όταν μιλάμε για συμφωνίες με την Βραζιλία. Όπως και να έχει, πρέπει να προστατέψουμε τα δάση. Ζητώ λοιπόν από τους συναδέλφους την ομάδα των Πρασίνων να συνεργαστούν επικοδημητικά και πρέπει θετικά να εμπλέξουμε τη Βραζιλία στο παιχνίδι. Σε αυτή τη συμφωνία ε, υπάρχει ένα κεφάλαιο για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη με την ενίσχυση εμπορικών επαφών. Ε, εκεί αναφέρεται συγκεκριμένα η προβληματική για το περιβάλλον, για τη βιώσιμη οικονομία ε, και την προστασία αυτών των στόχων. Νομίζω ότι αυτά πρέπει να μπαίνουν σε αυτό το θέμα. Η κυρία Ροτρίκες Πιενιέρο. Ευχαριστώ και συγχαρητήρια κύριε Χόγκαν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκπέμπει τριπλάσια ποσότητα ε, θερίων θερμοκηπίου από το Μερκοσούρα, αλλά είμαστε παγκόσμιοι ηγέτες ε, στην μετατροπή. Ε, έχουμε την Πράσινη Συμφωνία ε, για το 2050 για την οδετερότητα ως προς τον άνθρακα. Αυτό είναι καλό μεν, αλλά δεν είναι επαρκές. Θα πρέπει να δεσμευτούν όλοι και να συμμετέχουν όλοι. Η ατμόσφαιρα δεν γνωρίζει σύνορα. Γι' αυτό χρειάζεται να δώσουμε ιδιαίτερη σημασία στη συμφωνία με τη Μερκοσούρ με ένα φιλόδοξο κεφάλαιο για την ε, βιώσιμη ανάπτυξη που να είναι νομικά δεσμευτικό και να είναι ουσιαστικές οι δεσμεύσεις να εφαρμοστεί η Συμφωνία των Παρισίων για την κλιματική αλλαγή και να ε, υπάρχουν και κυρώσεις, να καταργηθούν οι προτιμήσεις αν δεν τηρούνται αυτά. Θα πρέπει η Βραζιλία να σταματήσει τη λαθρέα υλοτόμηση και αποψήλωση των δασών και να μειώσει κατά 43% μέχρι το 2030 ε, σε σχέση με το 2005 τις εκπομπές. Ε, είναι μία από τις λίγες χώρες αναπτυσσόμενες, τις μεγάλες που μπορεί να το κάνει. Θα πρέπει να εγγυηθούμε την ε, εφαρμογή της συμφωνίας, να επαγρυπνούμε και εδώ θα πρωταγωνιστήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Ζητώ συγγνώμη που σα διακόπτω, αλλά να ζητάτε τι ομάδε σα να σα δίνουν περισσότερο χρόνο. Δεν φταίω εγώ, τι να σα κάνω. Η επόμενη ομιλήτρια είναι η κυρία Σπυράκη, παρακαλώ, για ένα λεπτό κυρία πρόεδρε επίτροπε χόγκαν αναμφίβολα η συμφωνία ευρωπαϊκής ένωσης μερκοσουρ είναι σημαντική και είναι και προφανώς οικονομικά επωφελής αφού αφορά επτακόσια εκατομμύρια καταναλωτές και διαφυλάσσει τις προστατευόμενες ενδείξεις και μειώνει τους δασμούς. είναι όμως πρωτίστως μια συμφωνία εξαιρετικά προκλητική και ο βασικός λόγος που η συμφωνία αυτή είναι εξαιρετικά προκλητική δεν είναι άλλος από την περιβαλλοντική πιστοποίηση των προϊόντων που εισέρχονται στην ευρωπαϊκή ένωση. είναι απαραίτητο σήμερα επίτροπε χόγκαν να διαβεβαιώσετε τους πολίτες μας να διαβεβαιώσετε τους αγρότες της ευρωπαϊκής ένωσης τους αγρότες της ελλάδος ότι τα προϊόντα που θα έρχονται στην ευρωπαϊκή ένωση από τις χώρες της μερκοσουρ θα φέρουν περιβαλλοντική πιστοποίηση θα έχουν τους ίδιους κανόνες με τους κανόνες που έχει η ευρωπαϊκή ένωση η μερκοσουρ μπορεί ακόμα να αποτελέσει και έναν ισχυρό μοχλό πίεση. ώστε οι χώρες αυτές να μπορέσουν να μας ακολουθήσουν στον υψηλό στόχο του green deal για το. 2050. χιλιάδε πενήντα κυρίως όμως πρέπει να είμαστε ρεαλιστέ. ακούσαμε τις εξαγγελίε του επικεφαλής της βραζιλίας του προέδρου της βραζιλίας. αυτό σημαίνει ότι η